Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη χαρά να σας ενημερώνω, λέει ο πρόεδρος, ότι έχουμε μέλη ε, της Αντιπροσωπείας Εθνικής Συνέλευσης της Μαυριτανίας, το θεωρείο των επισήμων. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά. Ο κύριος Ελάρμπι, όλοι οι άλλοι ηγείται της αντιπροσωπείας και έχουν έρθει για να συναντηθούν με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλώς ορίσατε στις Βρυξέλλες και στο κοινοβούλιο μας. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Μαυριτανία είναι πάρα πολύ σημαντικέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι ο γόνιμος διάλογος μεταξύ των δύο συνελεύσεων μπορεί να συνεισφέρει και να ε, ενισχύσει τη σχέση μας, να συσφίξουμε τους δεσμούς μας και να βρούμε και νέα πεδία συνεργασίας Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαυριτανία. Καλώς ορίστε θερμά και πάλι.